Ιουνίου θα θεωρήσουμε ότι αυτή η ερμηνεία εγκρίνεται. Έχει ζητήσει κάποιο το λόγο, Κύριε Ομενερόιτε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη συνεδρίαση μιλήσαμε για τη Ρωσία. Είχαμε τότε ε, αποστείλει κάποια μηνύματα στον πρόεδρο Κομισιόν και Συμβουλίου για να μιλήσουν για τις ρωσικές εκλογές. Τώρα μάθαμε πως ε, αρνήθηκαν την εγγραφή σε ένα κόμμα στη Ρωσία. Ο ΑΣΕ ε, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα με την αποστολή παρατηρητών, οπότε θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να έχουμε μία δήλωση πρώτον για την κατάσταση στη Ρωσία και δεύτερον ε, να γίνει μία συζήτηση εδώ πέρα. Νομίζω πως είναι σωστό. Ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα θέλω να στηρίξω αυτό το αίτημα Επαφίεται βέβαια στην ε, διάσκεψη των ε, Πρόεδρων, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση ούτω ή άλλω ε, τον Ιούλιο που θα έρθει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος να γίνει μια σύντομη τοποθέτηση και συζήτηση. Ωραία, δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει ένα αίτημα, το σημειώνουμε και θα το διαβιβάσουμε στα αρμόδια όργανα. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Το οριστικό πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης ε, έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 9 Ιουνίου και σας έχει διανεμηθεί. Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να υποβάλω στην αίθουσα της ε, εξή τροποποίηση τη ημερήσια διάταξη. Την 5η, 23 Ιανουαρίου του 2011, η ψηφοφορία για την έκθεση Κάσλερ για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης αναβάλλεται για τη συνεδρίαση του Ιουλίου. Δεύτερον, η έκθεση του κυρίου Καταρέλα για τα ε, τρακτέρ τα οποία ε, διατίθεται στην αγοριά ε, βάσει του σχήματος ευελιξίας ε, θα περιληφθεί στην ψηφοφορία. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών σήμερα στις 4. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, επομένως οι τροποποίησεις αυτές εγκρίνονται. Κατόπιν, έχουν ζητηθεί εξή τροποποίησεις την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε η κοινή συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση να γίνει αμέσως μετά από τη συζήτηση για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πριν από την έκθεση ΝΤΕΣ για την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν θέλει κάποιος να μιλήσει. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει καμία δήλωση. Ωραία. Ψηφίζουμε απευθεία. Ποιο είναι υπέρ τη τροποποίηση. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Η ημερήσια διάταξη μένει ως έχει. Περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης. Η ομάδα της ενωτικη Αριστεράς ζήτησε να αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση η ψηφοφορία για τις εκθέσεις που περιλαμβάνονται στη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση. Οι διάφορες εκθέσεις που έχουμε στο θέμα αυτό. Δίνω το λόγο τον κύριο Κλούτε για να παρουσιάσει το αίτημά του. Παρακαλώ. Abstimmung, die Diskussion... Ζητάμε η ψηφοφορία για την οικονομική διακυβέρνηση να αναβληθεί όπως και η συζήτηση για τον Ιούλιο στην Ολομέλεια διότι έχουμε ακόμη συνεδριάσει του ΕΚΟΦΗΝ και ως εκ τούτου καθώς δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί απαιτούμε να έχουμε το δικαίωμα ως ευρωβουλευτές να εξετάσουμε τα, ε, όσα συζητηθήκαν. Δεν έχουν γίνει μεταφράσεις. Υπάρχει μεγάλη πίεση από πλευρά του Συμβουλίου να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα αλλά παρακαλώ τους συναδέλφους να αντισταθούν σε αυτές τις πιέσεις του Κοινοβουλίου και να υπερψηφίσουν την αναβολή της εξετάσεις και του αιτήματος. Ναι. Μπορώ να δώσω το λόγο σε έναν από τους εισηγητές ε, για να μιλήσει υπέρ και ε, σε κάποιον αγορητή για να ε, μιλήσει κατά του αιτήματο. Ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ του αιτήματο, ποιος είναι κατά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη χρειάζεται επιγόντως σοβαρή βάση για το ευρώ. Συζητάμε αυτό το πακέτο εδώ και μήνες και υπάρχει μια συμφωνία στο 98% με το Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να γίνει ψηφοφορία αύριο έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί δια της ψήφου στην Ολομέλεια και χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για να έχουμε τελική συμφωνία πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού για να υπάρχει μια δυνατή βάση για το ευρώ. Eh, Καλώς. Έχετε δικαίωμα να μιλήσετε υπέρ της πρότασης. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα σύνολο μέτρων στο οποίο έχουν παρισφρήσει λογικές τελευταία στιγμή σε επίπεδο Συμβουλίου. Δεν έχουν μεταφραστεί σε τις γλώσσες οι αλλαγές αυτές, υπάρχει μόνο στα αγγλικά το κείμενο. Αυτό τουλάχιστον μπόρεσα εγώ να δω και δεν είναι δυνατόν χάρη σε αυτό να αντιληφθούμε πλήρως το τι έχει συμβεί και τι έχει αποφασιστεί. Πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με μείζονο σημασία εξελίξει. Εξελίξει και γεγονότα που μπορεί να έχουν τεράστιε επιπτώσει για τι χώρε ε, και του λαού μα, δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Φερρυπίν στην Ελλάδα, φέρει Φερρυπίν στην Ιρλανδία. Και Φερρυπίν όπως φαίνεται και στην Πορτογαλία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το κείμενο αυτό να το χειριστούμε με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα και να στήσουμε την αναβολή για τον Ιούλιο της συζήτησης και ψηφοφορίας. Ωραία. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αίτημα. Συνεπώς έχει καθοριστεί η διάταξη. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο